Okay, dear colleagues, please may I ask you to take seat? Yeah, yourself. Yeah, yeah. And we are as well. <laughs> You are too. Yeah. Συνάδελφε, καθίστε. I... Καθίστε, λέει ο Πρόεδρος. Θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί μέσα σε διάταξη. Αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση, παρακαλώ, συναδέλφο, Λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμεθα τον Μάικλ Νούνεν, τον Ιρλανδό Υπουργό Οικονομικών. Για να έχουμε ένα διάλογο σε οικονομικά θέματα και ανταλλαγή απόψεων στην ε, Επιτροπή μας. Να δούμε πιο συγκεκριμένα την οικονομική συγκυρία στην Ιρλανδία, αλλά επίσης και τις ε, προοπτικές τη Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Καλώ ορίσατε, με μεγάλη μα χαρά σα υποδεχόμεθα και όπω γνωρίζετε, αφού η χώρα σα χτυπήθηκε πάρα πολύ σκληρά το 2010 από την χρηματοπιστωτική κρίση, η οικονομία σα ε, μετά ανέκαμψε εντυπωσιακά και το 2013 βγήκατε από το πρόγραμμα τη προσαρμογής της ε, Επιτροπή, της Τρόικα τέλος πάντων και ε, τον Ιούνιο δεν βγήκατε από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και έγινε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και έτσι προσθέμαστε πλήρως του 14 15 στην Ευρωζώνη και όπως ε, γνωρίζουμε τώρα έχουμε ε, υφηξημένε αβιότητες λόγω του Brexit οπότε αυτό είναι με καινούργια μεταβλητή φανεία αβέβαιότητα στο οικονομικό κλίμα, αλλά βέβαια και για την Ιρλανδία αυτό. Και σας δίνω κύριε Υπουργέ των Ευρωπαϊκών τον ε, λόγο για τις ε, παρατηρήσεις σας και κατόπιν θα ακολουθήσουν. Ερώτα Αντών Βουλευτέ. Αγαπητέ Ρομπέρτο, σας ευχαριστώ. Θέλω να σα ευχαριστήσω που με καλέσατε εδώ για να συζητήσουμε την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώ και την οικονομική χρηματοπιστωτική κατάσταση στην Ιρλανδία και πρέπει να σα πω ότι στην Ιρλανδία έχουμε κάνει πολύ δρόμο στην προσπάθειά μα να ανακάμψουμε τα τελευταία χρόνια όταν ανέλαβα το Μάρτιο του 2011 το έλλειμμα για το 10 ήταν 32% του ΑΕΠΑ και ακόμα και ξερώντας ε, τις ε, τραπεζικές συναλλαγές ε, εξακολουθούσαν να είναι 12% του ΑΕΠ. Σήμερα προβλέπουμε μόλις 0,4% του ΑΕΠ για το 2017. Το Μάρτιο του 2011 η Ιρλανδία δεν μπορούσε να δανειστεί στην αγορά, αλλά εξαρτώμασταν από το πρόγραμμα της Ένωση του Δενεστικού Ταμείου. Τα δεκαετή ομόλογα είχαν απόδοση 14% τον Ήλιο του 2011. Τον προηγούμενο όμω μήνα το Γραφείο Διαχείρισης Χρέους εξέδωσε δεκαετή ομόλογα 0,495 ανασέντα και τα ομόλογα του δημοσίου με αρνητικέ επιδόσει. Το Μάρτιο του 2011 η ανεργία ήδη ήταν 14,3% και έφτασε στα ανώτατα επίπεδα πάνω από 15% το Γενάρη του 2012, τώρα είναι 7,7%. Η Ιρλανδική οικονομία ανακάμπτει, η βιώσιμη ανάπτυξη προβλέπεται να επανέλθει. Προβλέπουμε ότι το ΕΠ θα ανεβεί κατά 4,2% το 16, κατά 3,5% το 17, Δύο εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στην Ιρλανδία και μπορεί να μην έχουμε φτάσει την ανώτατη τιμή του 2007. Προβλέπουμε όμως ότι θα έχουμε μια πλέον αύξηση κατά 43.000 ακόμη Ιρλανδούς μέχρι τα τέλη του 2017. Συνολικά για την Ευρωζώνη, τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του ΑΕΠ δείχνουν ότι η οικονομία στην Ευρωζώνη γενικά ανακάμπτει, βέβαια με μέτριο ρυθμό και αυτό στηρίχθηκε και από θετικέ εξελίξεις όπως είναι οι χαμηλέ τιμέ του πετρελαίου και μέχρι πρόσφατα η χαμηλή εξωτερική τιμή, ισοτιμία του ευρώ. Όμω φαίνεται ότι οι ουροί άνεμοι αυτοί σιγά σιγά θα ανακοπούν και έχουμε κίνδυνο λόγω τη επιβράδυνση τη οικονομίας και ανασφάλεια μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα. Έχουμε λοιπόν βραδεί ρυθμού ανάκαμψη και έχουμε και κλειοδοτήματα τη κρίση, όπω ε, χαμηλό πληθωρισμό, υψηλή ανεργία, επιπτώσει ε, του δημοψήφισματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε λοιπόν προκλήσει μπροστά μα και δεν μπορούμε να είμαστε αυτάρισκοι. Τα δημόσια οικονομικά της Ιρλανδίας, ενώ ήταν εντελώς ε, αβίωτη κατάσταση και βασιζόμαστε στο μνημόνιο ε, για την οικονομική υποστήριξη, έχουμε φτάσει σε βιωσιμότητα, έχουμε ξαναφτιάξει τη φορολογική μας βάση, επενδύουμε περισσότερο στις δημόσιες υπηρεσίες. Για το προπολογισμό, μάλλον φαίνεται ότι ε, το έλλειμμα το Γενικό Κρατικό Έλλειμμα θα είναι του ΑΕΠ για φέτος και θα συνεχιστεί πτωτικά για να φτάσει 0,4% το 2017. Επίση ε, θα έχουμε ένα δομικό έλλειμμα της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ. Με βάση αυτές τις ε, υποθέσεις ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε ένα μεσοπρόθεσμο φορολογικό στόχο του να έχουμε ε, έναν ισοσκελισμένο προπολογισμό μέχρι το 2018. Σε ό,τι αφορά τώρα το 76% του ΑΕΠ που ήταν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, νομίζω ότι θα είμαστε κάτω από το μεσόρο της Ένωσης, χαλαρά. Αυτό είναι σαφής ε, ένδειξη ότι έχουμε πρόοδο και για τα μέσα έως τα τέλη δεκαετίας του 20 θα έχουμε ένα χαμηλότερο στόχο, 45% του ΑΕΠΑ, για να οροφήσουμε περαιτέρω κραδασμούς ενδεχομένως. Έχουμε λοιπόν μια δημοσιονομική πλατφόρμα βιώσιμη, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις βιώσιμες δημόσιες υπηρεσίες για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, όπως γνωρίζετε ίσως, το δημοσιονομικό καθεστώς, το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθέτησης και ανάπτυξη, θα εξασφαλίσει τη βιώσιμη χρηματοδότηση των αξίσεων των δημόσιων δαπανών που θα αποσυνδεθούν από την εξάρτησή μας από τα κυκλικά έσοδα. Και είναι σχεδιασμένοι αυτοί οι κανόνε, ούτω ώστε η δημοσιονομική πολιτική να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Και είναι μια θετική αλλαγή. Η αντίδραση των αγορών στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ήταν θετική, αλλά αν θέλουμε να την υποστηρίξουμε θα πρέπει να μην είμαστε αυτάρισκοι, αλλά να παραμείνουμε πάρα πολύ σόφρονοι στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και να στραφούμε σε πολιτικές προσανατολισμένες στην ανταγωνιστικότητα. Τα στοιχεία του ΑΕΠ μπορεί να είναι ρευστά στην Ιρλανδία, το είδαμε και όταν αναγγείλαμε πριν από κάποιου μήνε ποσοστό ανάπτυξη 26% για το 2015. Αυτό το 26% το ποσοστό ήταν πολύ πιο πάνω από την προηγούμενη μα εκτίμηση, το 7,8% και επηρεάζεται, μάλλον στρεβλώνεται από τι πολυεθνικέ δραστηριότητε. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό και χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να τα αναφέρω αυτά, γιατί ξέρω σα ενδιαφέρει το θέμα. Λοιπόν, είχαμε επίτα ε, δελτίο αναθεώρηση λόγω των δραστηριοτήτων ενό μικρού μεγάλων πολυεθνικών. Και είναι και κάποιοι έκτακτοι φορεί ε, με έχουν όμως επηρεάσει την δραστηριότητα και της ελληνικής οικονομίας όπως ε, είναι η τερκή αναδιάρθρωση κειμένων περιουσιακών στοιχείων και κάποιες ανακατατάξεις των ισολογισμών. Πώς επηρεάζεται λοιπόν το ΑΕΠ είναι με το λεγόμενο contract manufacturing. Πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ιρλανδία ε, αναθέτουν παραγωγή ε, των προϊόντων σε τρίτες χώρες, σε εταιρείε τρίτων χωρών ε, και καταγράφονται παρόλα αυτά στο εμπορικό ισοζύγιο με βάση τα συμπεφωνημένα στατιστικά πρότυπα. Επίσης έχουμε την μετεγκατάσταση κάποιων πλώτων βεστιχνίας ή περιουσιακών αγαθών, αύξηση στα τέλη αεροδρομίου. Έχουμε διεθνές δραστηριότητες μίσθωσης ε, και τα λοιπά. Όλα αυτά δεν επηρεάζουν την πραγματική οικονομία. Δεν αλλάζει δηλαδή η κατάσταση πραγματικής οικονομίας, αλλά τα επίπεδα των δραστηριοτήτων επιτόπου. Μπορεί με όλα αυτά να βελτιώθηκαν οι επενδύσεις ε, και να έχουμε περισσότερες καθαρές εξαγωγές, όμως θα πρέπει να είμαστε ε, να έχουμε την επίγνωση του ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί και άμεσα πλούτος για τους Ελλανδούς πολίτες. Βλέπουμε όμως με άλλους ε, δείκτες ότι υπάρχει ανάκαμψη σταθερή. Ε, έχουμε δείκτες όπως είναι οι δαπάνες καταναλωτικές, οι φορολογικές τάσεις, η εξέλιξη στην αγορά εργασίας δείχνουν ότι τα βασικά οικονομικά μας μεγέθη είναι ισχυρά και θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε μια να βασίσουμε τις πολιτικέ μα στο πιο ρεαλιστικό ποσοστό ανάπτυξης γύρω στο 3,4%. Ε, μίλησα για τις, εξωτερικές, ε, τις εσωτερικές συγγνώμη, προκλήσεις. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για τις εξωτερικές προκλήσεις. Έχουμε το ε, δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είπα και στην αρχή ε, ότι πρόκειται για σημαντική πρόκληση. Για μας ένας πραγματικός κίνδυνος για την οικονομία, επειδή υπάρχουν στενές σχέσεις και εμπορικές μεταξύ άλλων. 16% περίπου των Ιρλανδικών εξαγωγών πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και το 40% των εξαγωγών των εταιριών μας. Ε, και σε αντάλλαγμα είμαστε ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγή ε, αγορά 1,2 δις ε, είναι οι ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών σε εβδομαδιαία βάση, 400.000 θέσεις εργασίας ε, μεταξύ των δύο νησών και πολύ περισσότερες θέσεις στην αυλισίδα εφοδιασμού. Υπάρχουν ανασφάλειες λόγω της, οικονομικής, της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου και έτσι θα μειωθεί η πρόβλεψή μας για ανάπτυξη του ΑΕΠ στο 3,5% για του χρόνου. Θα δούμε τι θα γίνει, θα συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορούμε αυτά να τα εκτιμήσουμε από τώρα, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε αρνητικές επιπτώσεις. Το καλύτερο αποτέλεσμα για την Ιρλανδία θα ήταν μια ε, σύνδεση, στενή σύνδεση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θέλουμε να έχουμε, ένα λεγόμενο, να έχουμε σύνορα ε, με τη Βόρεια Ιρλανδία τύχη ή αλλαγές που θα αναστρέψουν ε, την κοινή οικονομία. Θέλουμε να διατηρηθεί η κοινή ε, περιοχή και η διατήρηση της κοινή αγοράς εργασίας. 2,25 με 3,75 χαμηλότερο θα είναι το ΑΕΠ σε σχέση με αυτό που θα ήταν αν δεν είχε βγει η, το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση, αυτό σε 10 χρόνια. Θα όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα μελετήσουμε πολύ προσεκτικά και θα πρέπει να υιοθετήσουμε συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουμε κλάδους της οικονομίας και όπως είπα για να ελαχιστοποιήσουμε και τις επιπτώσεις μελλοντικών οικονομικών σοκ τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θα ήταν να διαχειριστούμε, να ελέγξουμε τα δημόσια οικονομικά με την δική μας δημοσιονομική διαδικασία, να συνεχίσουμε να είμαστε υπεύθυνοι. Να ακολουθούμε τη σόφρονα δημοσιονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα. Στον τελευταίο προπολογισμό στόχο ήταν η μείωση και η εξάλληψη του δημοσιονομικού ελλείμματο, ε, ο ισοσχελισμό του προπολογισμού του 2018 και από εκεί πέρα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα. Νομίζουμε ότι αυτή η σόφρονα προσέγγιση θα μα βοηθήσει στο μέλλον. Τώρα θέλω να μιλήσω για κάποια άλλα στοιχεία, ε, όπως είναι η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Τάτρα, ε, στη Σύνοδο Κορυφής, το Σαββατοκύριακο μίλησα για τους νοσομικούς κανόνες. Είπα ότι δέχομαι την αρχή των νοσομικών κανόνων, είναι κάτι αναγκαίο στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης για... για τις ε, στους φυσιολογικούς καιρούς που μπορούν να βοηθήσουν ε, στην αποτροπή προκυκλικών πολιτικών. Ε, είναι κάτι που το έχουμε αντιληφθεί στην Ιρλανδία και είμαστε η μόνη χώρα που είμαστε συμβαλόμενοι στη Συνθήκη σταθερότητα Συντονισμού και Διακυβέρνηση, στο λεγόμενο Δημοσιονομικό Σύμφωνο που έχουμε δημοψηφίσματα και γι' αυτό ε, και επειδή έχουμε αυτή τη δημοκρατική αντίληψη για τους κανόνες αυτούς και επειδή αντιλαμβανόμαστε τι προέκυψε από τις οικονομικές και δημοσιονομικές ε, κρίσεις, στηρίζονται αυτές οι πολιτικές. Το πολιτικό σύστημα έχει αντιληφθεί την ανάγκη να ρευστό πλαίσιο αυτών των δημοσιονομικών κανόνων και δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα σφάλματα του παρελθόντος. Η συνεννόηση είναι ότι θα βοηθήσει η συμμόρφωση προς τους ε, κανόνες αυτούς. Κάποιες φορές όμως ό,τι αφορά την εφαρμογή των δημοσιομικών κανόνων θεωρείται ότι δεν τα πηγαίνουμε καλά γιατί χρειάστηκε να προβούμε σε μια τεράστια δημοσιομική προσαρμογή από το 8 στο 15 δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαια αυτό κάτι δεδομένο και επίσης αυτή η έλλειψη διαφάνειας προβλεψιμότητας και η πολυπλοκότητα είναι χαρακτηριστικά των κανόν. Τι θέλω να πω. Νομίζω ότι πολύ συμφωνείτε με τις ανησυχίες μου ότι όπως έχουν συλληφθεί αυτοί οι κανόνες είναι άκρος πολύπλοκοι. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν κατανοητοί στον πληθυσμό και έτσι και των προτέρων δύσκολα μπορούμε να προβλέψουμε και την ε, αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες. Τεράστιο πρόβλημα αυτό για τους χαράκτες πολιτικής. Η διαθετική ισορροπία που είναι στο επίκεντρο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν γίνεται ευρέως κατανοητή, αλλά υπάρχει και μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει με την ασυνεπή μεταχείριση. Ιδίω ε, για τι μικρέ χώρε με λεφτό είναι ένα πρόβλημα στην Ιρλανδία. Εμεί προασπίζουμε του δημοσιονομικού κανόνε, εξηγούμε ότι είναι σημαντικό να του στηρούμε. Ωστόσο, είναι πιο δύσκολο να το υποστηρίξουμε αυτό όταν υπάρχουν και περισσότεροι που υποστηρίζουν δεν εφαρμόζονται με λογικό ή συνεπή τρόπο αυτοί οι κανόνε ή ότι ε, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, άλλα για τα μικρά και άλλα για τα μεγάλα κράτη-μέλη. Και είναι ένα θέμα που είναι φύγει βέστες χορδές για τα μικρά κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις των συμφώνων είναι καλοδεχούμενες. ευθυγραμμίζουν καλύτερα του κανόνε με τι οικονομικέ συνθήκε και δίνουν κάποια ευελιξία σε ό,τι αφορά τι επενδύσει και τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και πρέπει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Τώρα, οι έξι μήνε ε, τη Προεδρία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013 ε, έγιναν σε ένα διάστημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε την τραπεζική και χρηματοπιστωτική κρίση. Μεγάλη πρόοδος έγινε σε συνεργασία με όλους τους άλλους, με όλα τα άλλα θεσμικά όργανα και με τη δική σας επιτροπή. Από την πλευρά τώρα τραπεζών, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είχαμε δύσκολες μικροσκελείς διαβουλεύσεις, αλλά καταφέραμε να έχουμε μια πολιτική συμφωνία. Συμφωνήθηκαν τα βασικά για την Τραπεζική Ένωση, ε, το πακέτο για τις κεφαλικές απαιτήσεις, ο νέος οπτικός μηχανισμός, γενικές ε, ε, προσεγγίσεις του Συμβουλίου και τα λοιπά σε ό,τι αφορά την οδηγία για την καθάριση τραπεζών και άλλα στοιχεία του ενιαίου μηχανισμού εκαθάρισης έχουν ε, βελτιωθεί. Τώρα σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση έχουμε το δίπτυχο, τα μέτρα δηλαδή οικονομικής διακυβέρνησης που συμφωνήθηκαν επί της δικής μας προεδρίας και η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου εξαθολογίστηκε. Έχει γίνει βέβαια περαιτέρω δουλειά στον τομέα αυτό. Σίγουρα το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο, το πλαίσιο οικονομική διακυβέρνηση, ο ΝΕ, έχει υποστεί σημαντικέ αλλαγέ τα τελευταία χρόνια, που δεν ξέρουμε ακριβώ ακόμη τι επιπτώσει θα έχουν, ιδίω σε εθνικό επίπεδο. Τα περιθώρια ελιγμών για τα δημοσιονομικά ζητήματα είναι περιορισμένα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν όλοι μα προκλήσει και πρέπει να τα εξηγήσουμε όλα αυτά στου πολίτε μα. Ωστόσο, είμαστε συνεπεί ω στην άποψη ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην πλήρη αποτελεσματική εφαρμογή ενό ευρέω φάσματο οικονομικών και δημοσιονομικών μέτρων στον τομέα της διακυβέρνησης. Περιμένουμε και τη δημοσιοποίηση της Λευκής Βίβλου, την ε, άνοιξη από την Κομισιόν. Όμως εμείς θα ξεκολουθήσουμε να ε, προσπαθούμε να εκπλώσουμε το στόχο μας για απασχόληση, για ανάπτυξη Για να αντιμετωπίσουμε την ανεμική ανάπτυξη στην Ευρώπη θα πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις επενδύσεων, ε, προϋποθέσεις για θέσεις εργασίας. Ε, δεν μας βοηθήσουν οι δομές ευρωπαϊκές και διάφοροι τέτοιοι μηχανισμοί. Ε, θα πρέπει εκεί να εστιάσουμε. Επίσης, σήμερα συζητήσαμε στο ΕΚΟΦΗΝ διάφορα ζητήματα, όπως παρουσίαση κομισιών, ένα, ένα πακέτο για τον εταιρικό φόρο. 25 Οκτωβρίου δημοσιοποιήθηκε το σχετικό έγγραφο. Αυτό το πακέτο έχει ως βασικό θέμα την πρόταση για την κοινή νοποιημένη εταιρική φορολογική βάση. Πρόκειται ε, για μια πολύπλοκη πρόταση. Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικούς κανόνες για το φορολογικό εισόδημα, για τις απαλλαγές κτλ. Ξετάζουμε τώρα βέβαια, όπως και τα άλλα κράτη-μέλη, τις αναλυτικές ε, προτάσεις. Ό,τι αφορά τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, δεν θα σας εκπλήξω να σας πω η Ιρλανδία διαδραμάτισε έναν ενεργό ρόλο ε, στην προσπάθεια μεταρρύθμιση του Διεθνούς ε, Συστήματος Εταιρικών Φόρων. Εφαρμόζουμε από τους πρώτους ε, το σχέδιο τη ΟΣΑ, Base Erosion Profit Shifting, διάβρωση βάση και μετατόπιση κερδών. Συμμετέχουμε σε διάφορε σημαντικέ μεταρρυθμίσει. Έχουμε τι εκθέσει αναχώρα. Ένα σημαντικό μέσο και επίση στηρίζουμε τη φορολογική διαφάνεια και την διοικητική συνεργασία. Γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά θα μα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα παγκόσμια προβλήματα τη φόρο αποφυγή και του φορολογικού σχεδιασμού, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. ολοκληρώνοντα να πω δύο λόγια για την περίπτωση κρατικών ενισχύσεων. 30 Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα τη έρευνά τη σε σχέση με την Apple, τη φορολογική τη μεταχείριση στην Ιρλανδία. Εμεί από την αρχή είχαμε ξεκαθαρίσει τη θέση μα. Είχαμε πει ότι η κυβέρνηση διαφωνεί κάθετα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μας άφησε απόφαση άλλη επιλογή από το να ε, κάνουμε προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αύριο συγκεκριμένα. Και υπό το φως αυτό και επειδή ακόμα η νομική διαδικασία συνεχίζεται, ε, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω επ' αυτού. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και με τα χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις και τα σχόλια των μελών. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, ε, σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρουσιάσεις σας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Σας παρακαλώ λοιπόν το πολύ μισή λεπτό κάθε βουλευτής. Μπορκάρτ Χαρτμπάλτς. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε στον διάλογο μαζί μας σήμερα. Θα ξεκινήσω με τις μακροοικονομικές ε, προοπτικές ε, της χώρας σας. Η Κομισιόν ε, τον Σεπτέμβριο λέει πως έχετε εξαιρετικές επιδόσεις στην τις μεταρρυθμίσεις. Δεδομένης της εντυπωσιακής ανάκαμψής σας, ποια είναι τα πιο σημαντικά μαθήματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από την οικονομική προσαρμογή σας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλα κρατημέλη. Επίση, τι μπορεί να γίνει διαφορετικά και κατά την άποψή σας, ποια είναι τα σημαντικότερα μέτρα που έχετε λάβει μέχρι στιγμής. Αυτά για να έχετε και εσείς χρόνο να απαντήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το Μάρτιο του 2011 ε, βγήκαμε, ε, μπήκαμε στο πρόγραμμα. Το βασικότερο ήταν λοιπόν να πείσουμε και το κοινό και τους πολιτικούς να αγκαλιάσουμε θα έλεγα το πρόγραμμα γιατί ήταν πολύ δύσκολη η όρη και πολύ σκληρά τα μέτρα. Αφού έγινε όμως αυτό και το υιοθετήσαμε, επιμείναμε σε αυτό. Γιατί οπουδήποτε βέβαια ξεκινάει κανείς μια τέτοια διαδρομή και μετά παρεκκλίνει δεν θα βγει εκεί που θέλει. Οπότε ήταν σημαντικό να επιμείνουμε στο πρόγραμμα. Μετά είχαμε βέβαια τα μέτρα κάθε αυτά οι δημοσιονομικές διορθώσεις 20% περίπου των μισθών στην δημόσια υπηρεσία ένα μεγάλο επίδευμα και βεβαίω ε, σημαντικό κατόρθωμα της ε, κοινωνικής ε, συνεννόησης, συνεννόησης των κοινωνικών εταίρων. Επιπλέον, Λίγα πράγματα μπορούσαμε να κάνουμε στην πλευρά της ζήτησης ε, και ενσχυανά μοντέλα δεν θα λειτουργούσαν αν ήταν να αρχίζουμε να αυξάνουμε φόρους ε, οπότε επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ στις μεταρρυθμίσεις και στην πλευρά της προσφοράς. Ε, κατόπιν κάναμε ένα κάποιο είδους παράλληλο πρόγραμμα όπου ανά κλάδο προσπαθούσαμε να δούμε ποια ήταν τα προβλήματα σε κάθε κλάδο και να βρούμε κάποιες λύσεις. Παραδείγματος χάρη ο τουριστικός κλάδος δεν ήταν ανταγωνιστικός. Οπότε έπεσε ο ΦΠΑ από το 13% στο 9% ε, καταργήσαμε τον φόρο ταξιδίου, δώσαμε περισσότερα λεφτά στον Οργανισμό Τουρισμού για την προώθηση της Ιρλανδίας και γρήγορα άλλαξε η κατάσταση. Και έτσι διασώθηκε όχι μόνο ο τουρισμός, αλλά αυτή τη στιγμή ο τουρισμός φτάνει και στα λιγότερο πλούσια τμήματα της Ιρλανδίας που έχουν ωραία τοπία. Μετά επικεντρωθήκαμε στα ισχυρά μας σημεία, ο ισχυρός ήταν πάντα ε, μαζί με τη γεωργία σημαντικό κομμάτι της οικονομίας μας ε, και το είχαμε παραμελήσει οπότε επανήλθαμε σε αυτά. Θα είχαμε κάνει κάτι διαφορετικά, θα προσπάθησαμε να βρούμε ίσως περισσότερους πόρους ε, για κεφαλιακές επένδυσεις γιατί λόγω των δημοσιονομικών διορθώσεων μειώθηκαν οι προϋπολογισμοί και τώρα υπάρχει θα έλεγα έλλειψη υποδομών και οικονομικών και κοινωνικών και οι δημοσιονομικοί κανόνες ε, με περιορίζουν. Όσον αφορά την επένδυση στις απαραίτητες κοινωνικές ε, και οικονομικές υποδομές. Μάλιστα. Αναλύζει Ντόντ κατόπιν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια σας. Έχω τρεις γρήγορες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα αναφέρατε τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο για την Ιρλανδική οικονομία μετά το Brexit και μετά τις έρευνες του Υπουργείου Οικονομικών της Ιρλανδίας φαίνεται πως ε, κάνουμε περισσότερο εμπόριο με το Ενωμένο Βασίλειο και ε, προς τα εκεί μάλλον μας οθεί και η Ιρλανδική κυβέρνηση δηλαδή παρουσιάζει διαπραγματεύσεις σε ένα παιχνίδι όπου ό,τι κερδίζει ο ένας το χάνει ο άλλος ενώ τελικά αν έχουμε μια καλή συμφωνία θα αναγνωρίσουμε ακριβώς το ότι είμαστε αλληλένδετοι. Η Ιρλανδία είναι σε μια μοναδική θέση για να επηρεάσει την Βρετανική κυβέρνηση. Οπότε δεν ξέρω αν μπορείτε να τους παρακινήσετε να πάνε προς μια κατεύθυνση περισσότερη συνεργασίας κατόπιν. Ε, ο Πρωθυπουργός βεβαίως έχει ορίσει μια ομάδα συμβουλευτική με τα συνδικάτα, την κοινωνία των πολιτών, τι επιχειρήσει οπωσδήποτε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μα πείτε κάποια πράγματα, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο μετά το δημοψήφισμα. Και τέλο αναφέρατε την περίπτωση τη Apple. Αντιλαμβάνομαι πω βεβαίω βεβαίως δεν μπορείτε να μα πείτε τα πάντα, αλλά νομίζω πω αυτό δείχνει την ανάγκη να μεταρρυθμιστούν οι διεθνεί φορολογικοί κανόνες. Όπω ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει εδώ και καιρό την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Εγώ και ο συνάδελφος ο Νίτερ Μάρη το είχαμε ζητήσει. Είπατε ότι εξετάζετε τις ε, λεπτομέρειες της πρότασης της Κομισιόν για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Μπορείτε να μας πείτε αν την στηρίζετε επί της αρχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ενισχύουμε πάρα πολύ για το Brexit. Και έχουμε τρεις άξονες προβληματισμού για τις σχέσεις μας πρώτα πρώτα σαν ε, χώρα. Δεν θέλουμε τέλο πάντων να υπάρχουν κάποια διαπέραστα σύνορα μεταξύ ημών και της ε, <clears throat> Ευρωπαϊκή Ένωσης. Μιλάμε για 40 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Δουβλίνου. Οπότε και εμείς θέλουμε να συνεχιστεί αυτός ο κοινό χώρος για ταξίδι, κοινό εργασιακό χώρος. Αυτά υπάρχουν εκατοντάδες χρόνια πρώτα πρώτα έχουν ενσωματωθεί στο δικό μας δίκαιο και έχουμε συμφωνία με το νούμερο Βασίλειο το 1922 και τελικά όλα αυτά έχουν ενσωματωθεί επίση στην νομοθεσία μα. Επίση έχουμε κατά δεύτερον τι εμπορικέ ε, σχέσει, ακριβώ όπω είπα στην αρχή. Ε, είπαμε για δύο περίπου ε, δι αγαθά που διακινούνται και είμαστε αυτό θα είναι πρόβλημα αν βγει το νομοθεσμό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν μπορούμε κάτι να κάνουμε να επηρεάσουμε. Όσον αφορά τι ε, διμερεί εμπορικέ σχέσει. Προ το παρόν πάντω δεν μπορούμε να επηρεάσουμε και πάρα πολύ όσον αφορά τα τι διαπραγματεύονται και πώ διαμορφώνεται η κατάσταση μέσα από αυτέ τι διαπραγματεύσει με την ΕΕ. Αλλά συνεχίζουμε να προσπαθούμε, είμαστε σε συνεχή επαφή με του υπουργού. Αλλά και προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή ε, είχαν επαφή μαζί μας έγινε αυτή η επαφή είχαμε αυτή τη συνάντηση ε, σε ένα πύργο στο Δουβλίνο τελευταία φορά πάντως είχαμε κάποιο πρόβλημα στη συμμετοχή το DUP δεν συμμετέσχει ή την υπέρ του Brexit, όλα τα άλλα κόμματα της χώρας μας είναι κατά. Πάντως έχουμε πάρα πολλοί χειρούς δεσμούς σε διμερή βάση. Και για ιστορικούς και για άλλους λόγους. Ελπίζουμε επομένως ότι θα πάνε καλά οι σχέσεις μας και στη συνέχεια. Και διαπροσωπικές σχέσεις επίσης. Πάρα πολύ συχνά έχουμε στενές σχέσεις και πηγαίνουμε στο Belfast, στο Ulster επίσης θα γίνει κάποια συνάντηση μεταξύ των ε, αντιστοίχων ε, αρχών και κυβερνήσεων στα πλαίσια της Συμφωνίας Μεγάλης Παρασκευής. Και όσον αφορά την φορολογική βάση για τον εταιρικό φόρο, μας είπε μπράβο ο πρόεδρος του ΟΣΑ και θεωρείται πρωτοπόρα η νομοθεσία μας, η φορολογία. Ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια 2012 και 2013 και ο ίδιος έχω εμπλακεί με αυτό. Αλλά υπάρχει πρόβλημα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και έχουμε ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και ε, σωστά είπε ότι αυτό είναι θέμα προτεραιότητα η Σλοβακική Προεδρία. Θα πρέπει να είναι πιο εύρεθμη η επίλυση των διαφορών μεταξύ διαφορετικών κρατών στα φορολογικά ζητήματα. Επίσης, ο Επίτροπος Μοσκόβηση, απλώς διαδικασίας, χώρισε την κοινή βάση. Στον αφορά τη φορολογική βάση δηλαδή, λέμε καταρχήν ότι έτσι πρόκειται να στριμωχτούμε γιατί οι προτινόμενες εξαιρέσεις είναι ευρύτερε αυτών που εμείς είχαμε ρυθμίσει, είχαμε προβλέψει. Ελπίζουμε ότι πάντως θα βρούμε κάποιες συμβαστικές ρυθμίσεις πριν προκύψει η οριστική ρύθμιση. Κύριος Λούκε, θα μιλήσω γερμανικά. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας κατηγορεί ε, στην περίπτωση της Apple για παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Ρώτησα την κυρία Βεστάγκερ με βάση ποιο μέτρο σύγκρισης θεωρεί ότι ευνοήθηκε η Apple. Προς έκπληξή μου η κυρία Βεστάγκερ μου είπε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένα κάποια επιχείρηση με την οποία συνέκανε την Apple. Αν την περίπτωση Samsung. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου πείτε εσείς κάποια πράγματα. Κατά την άποψή σας η Samsung έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση με την Apple στην Ιρλανδία. Θα λέγατε δηλαδή ότι δεν υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ των δύο εταιριών. Και αν απαντήσετε με ναι, όπως υποθέτω, ε, να υποθέσω πως ε, και η Samsung έχει μία ανάλογη μεταχείριση. Δηλαδή υπήρξαν φορολογικές συνεννοήσεις και με την Samsung και η Samsung μπορεί να μεταφέρει τα κέρδη της σε μια έδρα, ένα head office όπου δεν φορολογούνται. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό του φόρου ε, του εταιρικού ε, φόρου τον οποίο πλήρωνε η Samsung στην Ιρλανδία 2003 μέχρι το 2012. Αν δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, ευχαριστώ και γραπτός δέχομαι κάποια απάντηση. Ευχαριστώ. Well, first of all, it's, uh, what you say is a true reflection. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο λέτε πραγματικά αντικατοπτρίζει την θέση της κυρίας Βεστάγκερ. Δεν υπάρχει κάποια σύγκριση, κάποιο μέτρο με, τον, με το οποίο να μπορούμε να συγκρίνουμε την φορολογική μεταχείριση της Apple. Και όπως λέτε, το κλειδί Ναι, όταν μιλάμε για κρατικές ενισχύσεις είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία να έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση από άλλες εταιρείες του ιδίου κλάδου. Και εδώ πέρα βεβαίως για φορολογικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο παράδειγμα. Και η γνωμοδότηση στην οποία βασίζεται η απόφαση αυτή είναι του 1991 και του 2007 και βεβαίω βασίζεται σε μια αρχή η οποία αναπτύχθηκε από τον ΩΣΑ την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας και τελικά αποκρισταλώθηκε σε κανόνες ε, μεταξύ 2010 και 2012. Η, θέση λοιπόν της Κομισιόν είναι πως υπάρχει κάποιος κανόνας που υπάρχει εντός των συνθήκων ο οποίος δεν αναφέρεται ρητός αν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι η Κομισιόν πέρασε 10-12 χρόνια συνεργαζόμενη με τον ΩΣΑ, για ποιο λόγο, για να αναπτύξει τον ίδιο κανόνα. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Τώρα μιλώντας για άλλες εταιρείε στην Ιρλανδία, τα φορολογικά ζητήματα είναι εμπιστευτικά και είναι ανεξάρτητος ο Επίτροπος της Φορολογίας, οπότε δεν, έχω, δεν έχω με μονομένη εταιρεία γιατί είναι κάτι το εμπιστευτικό. Αλλά οι φορολογικές αρχές μας έχουν πολύ καλή φήμη και η Επίτροπος Βεστάγκερ μου έχει πει ότι από όλους τους φακέλους που ζήτησε από την Ιρλανδία δεν υπάρχει καμιά άλλη περίπτωση που να εκρεμεί πέρα από την Apple για τα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων και ξέρετε πως ζήτησε αρκετούς φακέλους και συνεργαστήκαμε πλήρως με την αρχή ανταγωνισμού και δώσαμε όλα τα δεδομένα που μας ζητήθηκαν. Και αυτό περιλαμβάνει και τα δεδομένα και από τις φορολογικές αρχές, τον Επίτροπο Φορολογίας, στα οποία εγώ δεν έχω ως υπουργό πρόσβαση. Σε γενικές γραμμές όπως πολύ καλά ξέρετε, η φοροαποφυγή διεθνώς είναι συχνά αποτέλεσμα δραστηριοποίησης σε δύο δικαιοδοσίες όπου βλέπουν οι δικαιοβόροι ότι μπορούν να βρουν παραθυράκια στις νομοθεσίες δύο χωρών. Ε, μας δεν μας αρέσει τέτοια εκμετάλλευση και θα κλείσουμε όσο παραθυράκια μπορούμε και όπως είπα ξεκινήσαμε με τον ΩΣΑ, αλλά χωρίς διεθνή συνεργασία δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Εμείς φορολογούμε την Apple και όλους τους άλλους για τα κέρδη που έχουν στην Ιρλανδία, για τις δραστηριότητες τους στην Ιρλανδία. Αλλά αν βγάλω το τηλέφωνο μου εδώ αυτή τη στιγμή, βλέπετε πίσω γράφει σχεδιάστηκε στην Καλιφόρνια και κατασκευάστηκε στην Κίνα. Οπότε οι οικονομικές δραστηριότητες ε, δεν ε, λαμβάνουν χώρα στην ε, Ιρλανδία. Τώρα δεν ξέρω. Ε, μπορεί να μην, ε, να μην πλήρωσε αρκετό φόρο η Apple, αλλά δεν, είναι, δεν οφείλεται στην Ιρλανδία ο φόρος. Οφείλεται στις ε, διάφορες ακριβώς ασυνέπειες που υπάρχουν στις ΙΠΑ. Επίσης λέτε ότι δεν πληρώνουν φόρο για τα κέρδη τους στην Ιρλανδία, μα τα κέρδη δεν πάνε στην Ιρλανδία και βεβαίως ε, μην ξεχνάμε ότι και στις ΗΠΑ όταν επαναπατρίζουν κέρδη πληρώνουν 35% ε, εάν δείτε λοιπόν το φορολογικό βάρος σε σχέση με τα όσα πλήρωσαν είναι μεγάλο. Τώρα δεν ξέρω εγώ να σας πω πώς ακριβώς ε, λειτουργούν οι έφοροι παγκοσμίω, ε, εγώ βεβαίως συλλέγω τους φόρους για τις δραστηριότητες στην Ιρλανδία. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να μην υπάρχουν ασυνέπειες εντό του Ιρλανδικού δικαίου. Σα ευχαριστώ Μαριάν Χαρκίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και κύριε Υπουργέ, Έχουμε μια συγκεκριμένη ερώτηση που έχει να κάνει με το τι έγινε 2006 όσον αφορά την νομοθεσία για τους ε, γεωργούς όσο θα ξέρετε ότι έχω υποβάλει ένσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο επ' αυτού γιατί τώρα έχετε προβεί σε κάποιες ρυθμίσεις για την γεωργία μηχανισμό ούτω ώστε να εισπράξετε τον ε, ΦΠΑ με μία μέθοδο που είναι πάρα πολύ ζημιογόνα. Έτσι, όλος ο κλάδος της γεωργίας δεν μπορεί να είναι πια βιώσιμος. Επίσης, για πέστε μας, ε, ε, κάνατε μια τροπολογία στις 20 Οκτωβρίου φέτος όσον αφορά έναν ε, νόμο της οικονομικής πολιτικής, κάποια μέτρα, πάλι για την ίσπραξη του ΦΠΑ. Οπότε, για πέστε μας, πού θα ισχύσει αυτό το νομοσχέδιο. Θεωρείτε ότι η τροπολογία σας όσον αφορά την ίσπραξη του ΦΠΑ τι θα κάνει, δεν πρόκειται να αυξήσει τεχνητά τις τιμές των ε, ζωοτροφών. Έχουν προσφύγει οι γεωργοί και είπαμε ότι αυτού του είδους η επιστροφή αφορά τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Και όλο αυτό το κάναμε ούτω ώστε να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία. Εδώ και χρόνια ισχύει αυτό και έχει αποδώσει. Και οι επίτροποι ε, εσόδων έχουν λάβει την πρωτοβουλία αυτήν. Όχι εγώ. Είναι ανεξάρτητες αρχές. Και σε αυτό το ε, δημοσιονομικό νομοσχέδιο πρότεινε αυτή την τροπολογία για την ε, επιστροφή των χρημάτων και επίσης είχαμε κάποιες άλλες ρυθμίσεις για την ε, μη καταβολή του ΦΠΑ. Μην έχουμε έτσι, είπαμε, φοροδιαφύγη αφορά κυρίως την κτηνοτροφία. Έτσι υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε όποιους διαλέγουν να συμμορφωθούν προς αυτό το μέτρο. Τέλος πάντων έτσι, οι συμμορφούμενοι με τον νόμο δεν είναι πια οι χαμένοι όπως προηγουμένως. Το μέτρο θα ζητηθεί σε λίγο στο Κοινοβουλίο και ελπίζω ότι θα εγκριθεί. Ευχαριστώ Μακάρτη. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να ε, ξεκινήσουμε μια μακροοικονομική συζήτηση. Βέβαια, μιλήσατε για τη δημόσια υποστήριξη των δοσομικών κανόνων στην Ιρλανδία. Δεν ξέρω τελικά Μπαίνοντα στο αεροπλάνο, ήρθαμε από την ίδια χώρα και οι δύο εδώ. Άρχισα να αμφιβάλλω. Μιλήσατε για τη φορά που Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και εδώ πριν έρθετε συζητήσαμε τα περί των εγγράφων του Πανακά, Παναμά. Δυστυχώ, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη συνάντηση για το θέμα αυτό, αναφέρθηκε το όνομα της Ιρλανδίας και όχι θετικά. Και αυτό είναι λίγο ενοχλητικό. Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές συμφωνίες tax ruling, ε, τα έχουμε πει, ας πούμε κάτι διαφορετικό, είπατε ότι έχετε αναλάβει δράση σε αυτό το διπλό ελλανδικό καθεστώς, ε, το πολύ γνωστό, ε, διαβόητο. Και μιλήσατε για το 2014 και ότι από τον Ιανουάριο του 2015, θυμάμαι καλά, θα, σταδια, θα εξαβληφθεί σταδιακά, άρα οι εταιρείε αυτές θα θεωρούνται ότι ε, θα είναι φορολογικά υποκείμενες στην Ιρλανδία. Αφήνεται όμως μια, ε, ένα παραθυράκι για τις εταιρείε. Με κάποιο χρονικό ορίζοντα το 2020. Το Google δεν ξέρω τι θα προλάβει να κάνει μέχρι τότε. Είπαμε δεν θα συζητήσουμε τις μεμονωμένες ε, υποθέσεις, αλλά μπορεί σε αυτό το μεσοδιάστημα, το παραθυράκι που δίνεται μέχρι το 2020, να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους πολλές εταιρείες. Επίσης, φορολογικές συμφωνίες, μήπως ε, υπερβαίνουν ή καταργούν το εθνικό δίκαιο. Αν καταλαβαίνω καλά, α, τουλάχιστον αυτές τις συμφωνίες που διάβασα, θα μπορούσε να παραμείνει αυτό το ορλανδικό διπλό πρότυπο για χώρες όπως ε, ε, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ολλανδία, Βέλγιο, Μάλτα και κάποιες άλλες. Τι θέλω να σας ρωτήσω. Θα δεσμευτείτε ότι θα μειώσετε αυτό το παραθυράκι για τις επιχειρήσεις που ήδη έχει καταγραφεί ότι παραπέμπει το σύστημα. Και δεύτερον, θα επαναδιαπραγματευτείτε τις φορολογικές ε, αυτές συνθήκες, ε, συμφωνίες για να μπορούν να φορολογούνται εταιρείε μετά το 2020. Απάντηση. Όπως είπα, ε, προχωρούμε πάρα πολύ γρήγορα. Σίγουρα βοηθήθηκαν πολλές επιχειρήσεις λόγω της Ισλανδικής νομοθεσίας. Υπήρχε αυτό το φορολογικό, το double Irish που είπατε και μπορούσαν κάποιοι έξυπνοι φοροτεχνικοί να επιλέξουν ε, δύο διαφορετικές ή να επιλέξουν τη μία από την άλλη δικαιοδοσία και οι εταιρείε έτσι να διαφεύγουν τον φόρων που έπρεπε να καταβάλουν. Δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που συχνά μπερδεύουν κάποιοι. Είναι η φορολογική έδρα. Εκεί και σε σχέση και με το τι γίνεται σε άλλες δικαιοδοσίες υπήρχε μια περί κατάσταση. Εταιρείε, όχι ο ιδιώτε, ήταν απάτριδες για φορολογικούς λόγους. Δεν είχαν καταγραφεί κάπου. Όλα αυτά τα έχουμε βγάλει από το σύστημα. Σίγουρα. Έχουμε βάλει αυτή τη μεταβατική περίοδο, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Χρειάζεται και στο φορολογικό δίκαιο ασφάλεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα η δικαιοδοσία που μπορεί να αλλάξει τους κανόνες ε, ε, μέσα σε μια νύχτα για τον εταιρικό φόρο. Πάντα πρέπει να προειδοποιήσει. Αυτό κάναμε κι εμεί. Και είπαμε ότι από κάποια μέρα και μετά δεν θα μπορεί να ισχύει ότι ισχύει. Αλλά όσοι είχαν οργανωθεί, οι εταιρείε που είχαν οργανώσει τι εργασίε του και τι επιχειρήσει του με βάση τα όσα ίσχυαν, πρέπει να έχουν ένα περιθώριο χρονικό. Και ήδη πολλές, πάρα πολλές έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα συστήματά τους και προχωρούν στο νέο καθεστώς. Και αυτό ήδη πολύ πριν λήξει μεταβατική περίοδος. Σε ό,τι αφορά ε, τη δυσφήμιση που υφιστάμεθα ως Ιρλανδία, πράγματι ισχύει αυτό λόγω της υπόθεση της Apple, θα έλεγα. Και είναι και άδικο αυτό, θα έλεγα. Πολύ άδικο. και δεν θα πρέπει να παραποιούμε την ε, αλήθεια. Κάντε κι εσείς ό,τι μπορείτε για να μας υποστηρίξετε, να υποστηρίξετε φήμη της χώρας σας εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν απαντήσατε στο τελευταίο μου ερώτημα. Δεν ε, υπάρχει χρόνος. David Coburn. Thank you, Mr. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Σίγουρα, ο Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν αμοιβαίο συμφέρον υπάρχει ευημερία. Οικονομικό όφελο για του ε, Ιρλανδού. Αν υπάρχουν ανταγωνιστικοί εταιρικοί φόροι, υπάρχει. Αλλά υπάρχει αυτή η πρόταση για αυτή την ενοποιημένη εταιρική φορολογική βάση. Ξέραμε από τι χρηματοπιστωτικέ κρίσει ότι θα μπορούσε η Ιρλανδία να πληρώσει έτσι για τι απώλειε άλλων. Αν λοιπόν περάσει αυτή η πρόταση για την φορολογική βάση, πώς θα φροντίσει η Ιρλανδία να μην συγκεντρώνει φόρους μόνο και μόνο για να τους στέλνει στο εξωτερικό. Uh, uh, να απαντήσω στο τελευταίο ερώτημα που δεν απάντησε για τις φορολογικές συμφωνίες ότι περτερούν το εθνικό δικαίωμα. Αυτό ισχύει και είναι αρχή του διεθνούς δικαίου, άρα πρέπει να, στηρί... πρέπει να το εφαρμόσουμε το διεθνέ δίκαιο. Τώρα, για τον κύριο Κόμπεν, ξέρετε, είμαστε ένα μικρό κράτο και αγωνιζόμαστε με βάση την τιμή, την αξία, την ποιότητα και του φόρου, βέβαια. Έτσι έχουν τα πράγματα. Γιατί ο κόσμο είναι άκρο ανταγωνιστικό και έτσι δεξάγεται το εμπόριο. 12,5% είναι ο φορολογικός συντελεστής ε, και ίσχυε για πολύ καιρό αυτό. Στην Ηνωμένο Βασίλειο το ψηλό, ήταν πολύ ψηλότερο το ποσοστό. Αλλά ο Υπουργό Οικονομικών θα το μειώσει. Από 20, από, μάλλον θα το πάει σε 20, μετά 18 και κάτω ίσως πιο στο 15. αλλά είπε τώρα ότι ίσως δεν θα το κάνει, δεν θα φτάσει στο 15% κατά ανάγκη. Υπάρχει λοιπόν ανταγωνισμός φορολογικός σε όλη την Ευρώπη. Το πανεπιβεβαίωσε και η Κομισιόν πρόσφατα. Επιτρέπεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι ε, η φορολογική αρμοδιότητα εθνική. Και οι χώρες είναι ελεύθερες να ανταγωνίζονται με βάση φορολογικούς συντελεστές και αυτό θα κάνουμε και εμείς. Σημείωσα ότι στη συζήτηση για τον Brexit υπάρχουν κάποιε ενδείξει ότι ίσω το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρήσει σε χαμηλότερε χρονικού συντελεστέ. Εμεί ε, έχουμε προσελκύσει με μεγάλη επιτυχία μέσα στι ξένε επενδύσει. Αλλά η εταιρικοί φόροι και φορολογικοί συντελεστέ είναι μόνο ένα και όχι ο αποφασιστικό παράγοντα. Έχουμε όλο και πιο ε, μεγάλη μετακίνηση αν θέλετε, κινητικότητα επενδύσεων. Υπάρχουν πάντως καλοί λογιστές, φοροτεχνικοί, ε, προγραμματιστές, ε, υπολογιστέ και όλοι αυτοί. Επηρεάζουν επίσης. Εμείς στο μέλλον θα είμαστε μέλος της Ένωσης, θα είμαστε στην Ευρωζώνη και θα είμαστε τεχνή του δόρατος μιλάμε αγγλικά στην Ευρωζώνη. Και ίσως και αυτό να είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί μόνο εμείς και η Μάλτα θα είμαστε χώρες που θα έχουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επίσημη γλώσσα τα αγγλικά. Όταν ασκήσει το άρθρο 50 η Βρετανία. Το είπα ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για την ελλαδική οικονομία λόγω του Brexit. Δεν είναι όμως το πρόβλημα οι σχετικοί φορολογικοί συντελεστέ. αλλά η ανατροπή στα μοτίβα που είχαμε στο εμπόριο με τα γεωργοδιατροφικά προϊόντα κτλ. λοιπά, να γυρίσουμε πίσω στη θέση αναδίπλωσης αν χρειαστεί να διαπραγματευτεί τους εμπορικούς κανόνες ε, του ΕΒ θα έχουμε αλλαγές ε, με δασμούς, φορολογικά και όλα αυτά θα ε, χτυπήσουν άσχημα τις διμερείς εμπορικές μας σχέσεις. Δεν είναι το πρόβλημα όμως τόσο οι φορολογικοί συντελεστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Υπουργέ, η Ολλανδία, η Ολλανδία συγγνώμη, έχει στη δεκαετία του 10 και το 2014 60 εκατομμύρια σαν ενίσχυση και επίσης ε, από το 1973 έχει ε, ενισχυθεί από αυτά τα ταμεία. Κατά τη γνώμη σας τι θα γίνει το 2016. Πρόκειται η Ιρλανδία, η Ιρλανδία να βγει από τον έλεγχο και τι θα γίνει με την ελληνική από τους γείτονες. Ε, εσείς έχετε ελκύσει τις ε, πολυεθνικές με τους χαμηλούς φόρους και επίσης είχατε κάποιες ε, συμφωνίες ε, φορολογικές επιλήψιμες. Και καταφύγανε κάποιοι σε, σε φορολογικούς παραδείσους. Αυτό είναι εις βάρος των Ευρωπαίων εταίρων σας. Αυτών που προηγουμένως σας βοήθησαν. Μιλάμε για 13 δις ευρώ. Αυτά που η Apple έπρεπε να καταβάλει δεν τα εισπράξατε. Έτσι δεν είχαμε την δίκαιη κατανομή αυτών των πόρων. Αλλού όμως πληρώνονται αυτοί οι φόροι. Πρόκειται να συνεργαστείτε πάνω σε αυτό περισσότερο από ό,τι σήμερα. Να δεχτείτε να εισπράξετε αυτό το πρόστιμο. Εάν ναι, πότε θα το κάνετε αυτό και πώς. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Βεβαίω και εκτιμούμε την βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων και του Νομισματικού Ταμείου. Βεβαίω και με την ύφεση ήμασταν στα πρόθυρα της πτώχευσης και αναλάβαμε τις ευθύνες μας για το ότι φτάσαμε εκεί, οπότε και είμαστε ευγνώμονες και προς τους Ευρωπαίους εταίρους και προς το νομισματικό ταμείο μας έδωσε αυτά τα χρήματα. Έτσι προχωρήσαμε και κάναμε τις αναγκαίες προσαρμογές. Φυσικά δεν θα μπορούσαν αυτά να γίνουν από το βράδυ στο πρωί, ήταν καταστροφικό. Δεν μπορούσαμε να βγούμε τις αγορές. στην Ευρωζώνη. Βοηθηθήκαμε. Βέβαια αυτό είναι και υπέρ της Ευρωζώνης και των εταίρων μας, γιατί αν δεν μας βοηθούσαν, τότε έτσι που ήταν η Πορτογαλία, Ισπανία, η Ελλάδα, ε, θα έφερναν την κατάρτιση της Ευρωζώνης. Φυσικά και πρόκειται να πληρωθούν όσα πρέπει να πληρωθούν 22 δις προς το νομισματικό ταμείο τέσσερα, δις που μπορούμε να κρατήσουμε και έχουμε τώρα την υποπτία τους για να πληρώσουμε τελικά τα 18 από τα 22 και το τελευταίο ευρώ με το οποίο μας ενίσχυσαν οι Ευρωπαίοι εταιροί όπως προβλέπουν αυτά τα δάνεια σύμφωνα και με τους προβλεπόμενους τόκους. Κανείς δεν θα είναι φτωχότερος λόγω της κατάσταση, ε, κατάστασης της διαδρομής της Κατά δεύτερο λόγο δεν έχει επιβληθεί στην Apple κάποιο πρόστιμο. Δεν υπήρξαν αποδείξεις παρόμοιες δραστηριότητες. Απλώς απόφαση ότι δεν κατέβαλε η Apple τους δέοντες φόρους στην χώρα. Οπότε αυτά τα, τα χρηστούμενα θα αναζητηθούν. Εμείς, για αυτό το λόγο που προανέφερα, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει οφείλη της Apple προς την Ιρλανδία. Κατέβαλαν ότι όφυλαν. στο Κόρκ απασχολούν 6.000 Ιρλανδούς, καταβάλλονται εκεί ότι οφείλεται οι φόροι. Δεν ξέρω αλλού τι γίνεται. Εμεί κάνουμε ό,τι λέει ο ΣΑ. Όπου παράγεται κάποιο πλούτος, όπου αποκομίζεται κάποιο κέρδος, εκεί θα πρέπει να καταβάλλεται ο φόρος. Και όχι αλλού. Δεν φταίμε εμείς για το ότι υπάρχουν κάποιο είδους παραθυράκια του διεθνούς φορολογικού συστήματος στο οποίο έχουν κάποιοι έξυπνοι δικηγόροι. Εμείς θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις αθήνες πρακτικές. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση από κοντά μόνο από όταν γίναμε κυβέρνηση και συνεχίζουμε. Γιατί να πληρώνουν παραπάνω φόρους οι εταιρείε εκεί που δημιουργούν τα κέρδη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα μπορούσε κανείς να αλλάξει το διεθνές δίκαιο, όχι το κρατικό δίκαιο, ούτως ώστε να μην υπάρχει φοροδιαφυγή. Νομίζω ότι όπως πάμε θα τα καταφέρουμε. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Υπό την αιγίδα και, την, ε, και του όσα. Σας ευχαριστώ. Πρέπει τώρα να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις γιατί ο χρόνος τελειώνει. Brian Hayes. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Γνωρίζω πως ε, για εμάς και στην Ιρλανδία ο ρόλος σας ε, αναγνωρίζεται στην αποκατάσταση των οικονομικών της Ιλλανδίας. Να θέσω μια ερώτηση. Πριν μιλήσατε για το ότι το καλύτερο αποτέλεσμα για το Brexit θα είναι να είναι κοντά το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναρωτιέμαι, μιλάμε για πολλές δουλειές στην περιφερειά μου, το 1 τρίτο του Ιρλανδικού ΑΕΠ που σχετίζεται με τη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπετε λοιπόν κάποια δυνατότητα να διατηρηθεί η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο και τι είναι άποψη έχετε για τη δήλωση που έγινε πρόσφατα από Γερμανούς εξωματούχους ότι αν διατηρήσει η Μεγάλη Βρετανία τα δικαιώματα πώληση των ε, χρηματοπιστωτικών τη υπηρεσιών θα πρέπει να δεχτεί τι βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε, ε, είναι λίγο άχαρο να παίρνει κανείς το λόγο τελευταίος, αλλά τέλος πάντων. Θα ήθελα να μου πείτε το εξή. Μπορώ να τα πω στη γλώσσα μου, υπάρχει ερμηνεία. Ναι, υπάρχει βεβαίω. Μπερβάν, ε, θα είμαι σύντομο, δεν πειράζει. Ε, Έλεγα λοιπόν και από περίεργεια το ρωτάω, ποια είναι τα τρία σημαντικότερα πράγματα που θα κάνατε για να αποφύγετε να μετατοπιστούν τα κέρδη σε άλλο κράτος μέλος. Δηλαδή πώς θα αποφύγουμε όλα αυτά τα μοτίβα, όλα αυτά τα, τα, μέτρα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, που τα λέμε σήμερα. Τι θα θέλατε να κάνετε για να καταπολεμήσετε καλύτερα την φόρο αποφύγη, για να το πω αλλιώς, γιατί εμείς έχουμε καθήκον να πετύχουμε αυτούς τους στόχους 265 δισεκατομμύρια είναι τα έσοδα, ενώ έχουμε μαύρα διαφυγόντα κέρδη 2-3. Τι μπορείτε να κάνετε και εσείς για να πάψουν αυτές οι διαρροές κεφαλαίων. Ιβάνα Thank you, Καλώς ήρθατε κύριε, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και που ακούμε και αυτά που λέτε. Γιατί είστε πολύ έμπειρος και τα καταφέρατε πολύ καλά στην Ιρλανδία, πιστεύω. Την... Βλέπουμε την χώρα σας ως ένα καλό παράδειγμα, εμείς στην Κροατία, ότι έχει εφαρμόσει ένα καλό μείγμα πολιτικών για την τόνωση της οικονομίας. Έχω ένα ερώτημα σε σχέση με αυτό που και εσείς υπογραμμίσατε μεταξύ άλλων, ότι δηλαδή θα πρέπει να αυξηθούν οι κεφαλικές επενδύσεις, και μιλήσατε για κοινωνικέ και οικονομικές υποδομές κυρίω και είδα και στην έκθεση τη Κομισιόν ότι ειδικά αναφέρονται στην υδροδότηση, στέγαση, μεταφορές και σχετικά. Πώς λοιπόν βλέπετε το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων βοηθάει. Είναι ένα καλό εργαλείο. Θα τονώσει τις κεφαλαϊκές επενδύσεις, θα στηρίξει τις αλλαγές στην Ιρλανδία. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις ε, σε ό,τι αφορά και ένα μεγάλο ποσοστό των ε, τοξικών δανείων, των μη ε, αποπληρούμενων, εξυπηρετούμενων, συγγνώμη. Ο Πέτερ Ζήμων. Γεια, yeah, Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι η φορολογική νομοθεσία στην Ιρλανδία ε, η οποία πετέλεσε αντικείμενο κριτικής όπως το Double Iris έχει αλλάξει σε πολλά σημεία και είπατε πως υπάρχει διεθνής νομοθεσία η οποία ε, οδηγεί στο ότι εσείς ε, ε, συλλέγετε τους ε, Ιρλανδικούς φόρους, ε, αλλά όλοι οι υπόλοιποι σας ξεφεύγουν. Κάτι το οποίο βέβαια δεν ικανοποιεί τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνουν αυτά στην Ιρλανδία, την χώρα ακριβώς η οποία δέχτηκε και δισεκατομμύρια σε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ψηφοφόροι μου είπαν αφού δίνουμε βοήθεια στην ε, Ιρλανδία πρέπει να αλλάξει κάτι γιατί θεωρούν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια χώρα η οποία ζει εις βάρος των άλλων. Τώρα με την περίπτωση Apple πραγματικά δεν είναι κατανοητό πως μια χώρα η οποία ωφελήθηκε από την αλληλεγγύη των άλλων έχει ένα σύστημα το οποίο είναι εις βάρος όλων των υπολείπων. Μπορεί να είναι νόμιμο αλλά ε, όπως το βλέπουν οι ψηφοφόροι μου είναι 100% αθέμητο. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ Φουβίο Μαρτουσέλου. Για διευκρινίστε μου για τις δύο ερωτήσεις σχέση με την Apple. Αν λάβουμε υπόψη το τι έγινε. Γιατί δημιούργησε πολλές δυσκολίες σε αυτή την κατάσταση για τις επιχειρήσεις ε, που προχώρησαν από την Υπηρετική Ευρώπη και δρούν στην Ιρλανδία. Τι έγινε με τα έσοδα και τα εισοδήματα. Ε, τι γίνεται με τις ε, διμερείς συμφωνίε που έχετε με άλλες χώρες. Για πέστε μας. Θα αλλάξετε το φορολογικό σύστημα. Τι γίνεται επίσης με τις αμερικανικές εταιρείες που δρούν στην Ιρλανδία και ωφελούνται από το Double Irish. Μάλιστα, ο κύριο Τσόλτος. Και καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Πώς πρέπει να σας πάρουν σοβαρά οι Ευρωπαίοι σας όταν προσπαθείτε να μας πείσετε ότι ιστορικά και γεωγραφικά η Ιρλανδία ε, είναι τόπος όπου εξυπηρετεί τις φέρετε των εταιριών όταν έχετε αυτού του είδους την νομοθεσία. Και τι γίνεται με το ότι προσπαθείτε με τους συντελεστές να ξεπεράσετε τα δημοσιομικά προβλήματα και με τις φορολογικές συμφωνίες. Minister. Well, Σας ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας. Η ερώτηση του Brian Hayes για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικός. Εκτείνεται και εκτός Δουβλίνου. Είναι μια μικρή οικονομία, δηλαδή 38.000 θέσεις εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμάς. Υπάρχουν κάποια ωφέλη από το Brexit, γιατί όπως ε, το City του Λονδίνου πλέον δεν θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εταιρείε στο City που αναζητούν εναλλακτικέ ε, για να εγκατασταθούν και εναλλακτικέ είναι ευρωπαϊκές πόλει ε, μεταξύ των οποίων και το Δουβλίνο έχουμε, δεχόμαστε ήδη πολλά ερωτήματα και για πολύ σημαντικές εταιρείε από το City του Λονδίνου που προσπαθούν να πληροφορηθούν ποιο θα είναι το καθώς βέβαια εξετάζουν και το Άμστερνταμ, το Λουξεμβούργο, το Παρίσι, τη Φραγκφουρτή. Υπάρχουν επίσης εταιρείε από τις ΗΠΑ οι οποίες ε, πριν από το Brexit θα κοίταγαν το Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα εξετάζουν την Ιρλανδία. Χωρίς βεβαίως να ξέρουμε αυτή τη στιγμή το τι θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, μάλλον θα έλεγα ότι λαμβάνουν τα μέτρα τους παρά κάτι πιο συγκεκριμένο. Με ρωτήσατε για τρία βήματα που θα έπρεπε να αποφευχθούν. Η φοροδιαφύγη και η φοροαποφυγή. Το πρώτο βήμα είναι να εφαρμόσουμε τα συμφωνημένα. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας νέος κανόνας στην Ευρώπη, να εφαρμόζουμε τα συμφωνημένα, γιατί συμφωνούμε περισσότερα από όσα εφαρμόζουμε και αν ε, τα συμφωνημένα σε επίπεδο ΩΣΑ τα εφαρμόζαμε διεθνώς ε, το, αυτό θα έκανε τώρα μεγάλη διαφορά σε φορά φυγή και φορά φυγή δεύτερον αν οι νόμοι της κάθε χώρας αντικατόπτρισαν ε, την πραγματικότητα ο φόρος θα αφιλόταν και θα πλήρωνόταν εκεί όπου λαμβάνει η χώρα η οικονομική δραστηριότητα και όχι εκεί όπου βγάζαμε δίσκο ε, και βεβαίως έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος ε, στον ΩΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων αρχών. Αλλά αυτό το οποίο θα τόνιζα είναι ότι στην Ευρώπη και στο επίπεδο του ΩΣΑ συνεχώς ε, αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις οι οποίες δεν τηρούμε. Και αν το κάνουμε αυτό, δηλαδή τηρούσαμε τις δεσμεύσεις μας ε, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης αναφέρατε με ρώτησα κάποιος για τις ε, κεφαλαιακές επενδύσεις και το σχέδιο Juncker. Πάρα πολύ καλό, αλλά έχουμε περιορισμού στην Ιρλανδία λόγω των δημοσιονομικών κανόνων που περιορίζουν την ικανότητά μας για δαπάνες πέρα από ορισμένες παραμετρούς. Έχει όμως σημειωθεί πρόοδος ε, με τις ε, ΣΔΙΤ ε, και με άλλους κανόνες και, και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Και καθώς πάμε προς μια θέση ίσως και λιμένου προϋπολογισμού θα έχουμε περισσότερα περιθώρια για να χρησιμοποιήσουμε πόρους για τομεακές ε, μεταρρυθμίσεις. Ε, υποστηρίζουμε λοιπόν το σχέδιο Juncker και έχει πολλά ωφέλη νομίζω, θα έχουμε πολλά ωφέλη στο μέλλον. Ο κύριος Φέρμπερ ρώτησε για το γιατί μόνο στην Ιρλανδία, μα δεν είναι μόνο η Ιρλανδία. Αν δείτε το τι κάνουν οι δικηγόροι που ασχολούνται με τα φορολογικά, υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη. Δεν θα πω ονόματα, όπου γίνονται αυτές οι διευθετήσεις. Η Ιρλανδία φαίνεται γιατί ήμασταν πολύ επιτυχείς στον να ε, προσελκύουμε άμεσες ξένες επενδύσεις. Ε, είναι μια εύκολη χώρα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, μιλάμε αγγλικά, είμαστε στην Ευρωζώνη, έρχονται πολλές από αυτές ε, και στείλουν έδρα στην Ευρώπη, στην Ιρλανδία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο εικονικό. Υπάρχει πραγματική δραστηριότητα. Η Apple έχει 6.000 υπαλλήλους στην Ιρλανδία. Άλλα είναι τα ζητήματα, οι άλλες δραστηριότητες που δεν είναι φορολογητές στην Ιρλανδία. Ο κ. Ματιτσέλο νομίζω είπε κάτι παρόμοιο. Και νομίζω πως αν κάναμε όλοι ό,τι μπορούμε Αυτά ακριβώς τα ζητήματα φοροαποφυγής δεν θα τα είχαμε. Το θέμα για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων το έθεσα, το απάντησα ήδη. Και συνεργάζομαι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας και τον Επίτροπο Μοσκοβισή και έχω τονίσει πως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην υβρεδική κατάσταση που παρουσιάζεται στο έγγραφο αυτό και στο ψήφισμα για τις ε, φορολογικές διαφορές μεταξύ διαφόρων ε, δικαιοδοσιών. Δεν εργό λοιπόν, έχουν παρέλθει αυτές οι εποχές για την Ιρλανδία. Συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε την καλύτερη λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, χρήσιμη και ενδιαφέρουσα η επαφή μας. Βεβαίως ε, έχουμε συζητήσει τα ζητήματα φορολογίας και τώρα έχουμε και μια θετική πτυχή ε, με τις δεσμεύσεις που αναφέρατε. Μας εξηγήσατε λοιπόν τις αρχές και την στήριξη για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων. και βεβαίως αυτά θα μας απασχολήσουν στο μέλλον μαζί με το Brexit και άλλα θέματα. Θα είμαστε λοιπόν σε στενή επαφή. Ο κύριος Ντεγκίντος θα έρθει για τον επόμενο διάλογο το επόμενο ζήτημα μας. Λοιπόν, διάλειμμα.